την επόμενη συνεισμένη τώρα, το Ευρωπαϊκό Λεκό Κόμμα έχει έτοιμα σε σχέση με τον κύριο Φίσα, ο οποίος θέλουμε να ενταθεί στην προσωπία με την ε, σχέση με την Παλαιστίνη και να υπάρξει αντικατάσταση από, τον κύριο, την κυρία Ερμήνια. Οπότε θα γίνει έτσι σε αυτή την αλλαγή του ενός